Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Έχουμε τις ψηφοφορίες. Ε, ε, Θα ήθελα να πω στην αρχή ότι θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ, ετοιμαστείτε για αυτή τη δοκιμαστική ψηφοφορία, πολύ σημαντική. Καθίστε και πάψτε τις συζητήσεις, διότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την δοκιμαστική ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι για τις διακοπές. Απαντήστε παρακαλώ. Είστε έτοιμοι για διακοπές. Άρχεται η ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, συγγνώμη που είμαι γεννής, αλλά παρακαλώ σταματήστε να συνομιλείτε μεταξύ σας και αρχίστε να απαντάτε το ερώτημα που σας έθεσα. Λοιπόν, ωραία, πέρασε ψηφοφορίας. Επόμενο. Έχει γίνει μια μικρή αλλαγή στην σειρά των εκθέσεων που θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε πρώτα τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Συνάλλητος Αγγέλικα Νίμπλερ το ζήτησε γιατί πρέπει να μας εγκαταλείψει. Οπότε αλλάζουμε πρώτα το 5 μετά το 4. Δεν νομίζω ότι σας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Άρα ξεκινάμε με το σημείο 5 οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Κύριε Αγγέλη Καρνίμπλερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να καθυστερήσω την ψηφοφορία. Απλώς δράτω με τις ευκαιρίες για να απευθυνθώ σε όλους τους κοιόδης ηγητές και να τους ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για την έκθεση αυτή. Ξέρετε ότι υποβλήθησαν πολλές τροπολογίες, αλλά καταφέραμε στο τέλος να τις βρέψουμε όλες προς την διακατεύθυνση και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε σήμερα μέσω της έγκρισης έκθεσης αυτής να στείλουμε ένα χειρόθετικό μήνυμα προς όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν σε όλη αυτή την εργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τροπολογίες και για τις συμβαστικές τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε. Όλοι λοιπόν ε, συμβάλλατε και γι' αυτό θα ήθελα για άλλη μια φορά να σε ευχαριστώ για την αγαστή συνεργασία. Να πω το εξή ότι υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Ίσως ε, ο κύριος Πρόεδρος μπορεί μετά να μου δώσει τη δυνατότητα ε, πριν ψηφίσουμε για αυτή την προφορική τροπολογία να λάβω και πάλι το λόγο. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Συμβιβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67, 75 και 79. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 69. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Η 68 καταπίπτει και ψηφίζουμε είναι 69. Τροπολογία 69. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλ 25. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία. Παρακαλώ. Τροπολογία 72, 71, 73, 74. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβα... Μάλλον τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές να ελέγξουμε. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 97. Πέραση της ψηφοφορίας. Α, συγγνώμη. Είναι υπεράριθμη η του ΕΛΚ. Ένας παραπάνω. Εντάξει τώρα. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 98. Κύριε Νίμπλερ, εδώ έχει μια προφορική τροπολογία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν την εξής προφορική τροπολογία για την ε, τροπολογία 98 και παραθέτω καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της ε, ε, τα, τους, τα μέτρα που ισχύουν για τους αποδέκτες και εδώ έρχεται η προσθήκη με οικογενειακές επιχειρήσεις. Τέλος της αλλαγής. Το οικογενειακές επιχειρήσεις δηλαδή είναι η προσθήκη. Το ερώτημά μου είναι υπάρχει ένσταση. Αν κάποιος δεν θέλει την προφορική τροπολογία πρέπει να εγερθεί. Ουδής. Μάλιστα. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 98 με την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 137 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή τροπολογία 100 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 100. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 και 116 από κοινού. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. 112 και 116. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν οι τροπολογίες αυτές. Συμβιβαστική 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 110 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 9 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 της έμπλ υπέρ κατά αποχές και αυτή γίνεται δεκτή. Τροπολογία 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 138 ε, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 141 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 142 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 143 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά. Συγγνώμη, θα ελέγξουμε την 147 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν το συγγνώμη, αλλά δεν σηκώνατε τα χέρια. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια καλά. 149 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη 3, πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Από την τροπολογία 3 της Επιτροπής Απασχόλησης. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 189 υπέρ Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 189 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΦΑΜ 1. Τροπολογία Επιτροπή Γενικών. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ΦΑΜ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. ΦΑΜ 13 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τη 13 από την Επιτροπή Γυναικών. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβεβαστική 13 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τροπολογία 190 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 210. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα τη 210 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 15. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 7. Τροπολογία 7. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Κάποιος άλλαξε γνώμη. Το είδα. Γιατί πριν ήταν πολύ αμφιρό από 50-51, τώρα είναι μεγάλη διάφορα. Άρα να ελέγχω κάθε φορά. Λοιπόν, τροπολογία, όχι 8. Ναι, τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24, 25, από κοινού, υπέρ, κατά. Μάλλον απορρίπτονται, αλλά ας ελέγξουμε. 24 και 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. ψηφοφορία. 23 υπέρ. Μάλλον δεν ψήφισε κανεί. Λοιπόν, 23 ψήφι υπέρ. Κατά. Ποχέ. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Νομίζω. Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε καλύτερα την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Παραπορήθηκε. το πέτυχα. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά αποχές. Ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. Τροπολία 36 υπέρ. Κατά. Ξαναρχίζω. 36 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. MPG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. N νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 έμπλη πάντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε έμπλη 27. 27. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 28. Έγινε δεκτή 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Ελέγχουμε την 28. Λυπούμε. 28 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Καλά το είδαμε εμείς. Φαμ δι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Λυπούμε, αλλά δεν μπορώ να προβλέψω το αποτέλεσμα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε, θεούλη μου. Φαμ ε υπέρ. Κατά. ΑΠΟΧΕΣ, Απορρίφθηκε. G υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την G, Επιτροπή Γυναικών. Υπεράριθμη από το έλκα ένας παραπάνω. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. H. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Άι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε, λυπούμε, την K, Επιτροπή Γυναικών, ΦΑΜ K. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. ΦΑΜ 5, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 19 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα ονομαστικά μπορούμε να πούμε σχεδόν για το σύνολο της τελική ψηφοφορία άρχεται One PP. too many. Ένας υπεράρθρος από το ΕΛΚ Μήπως είναι η Αγγέλικα Νίμπλερ. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας. 48 ψήφοι υπέρ, συγχαρητήρια. Έχουμε το αποτέλεσμα λοιπόν. Συγχαρητήρια Αγγέλικα, περνάμε στο επόμενο σημείο. <laughs> Okay. Uh, the next is on the Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Γαλάζια οικονομία. Ο κύριος Φερέιρα είναι ο συγηγητής για την έκθεση αυτήν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά για την 93 ψηφίζουμε. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 121 άρχιτη ψηφοφορία πέρας Ισοψηφία και απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται, με συγχωρείτε, 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18, συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 152 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 και για την τροπολογία αυτή ο κύριος Φερέιρα θα ήθελε να μας πει κάτι. Παρακαλώ κύριε Φερέιρα έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπήρξε μία παρανόηση την οποία θελήσαμε να αποκαταστήσουμε μέσω μίας διευκρίνησης. Γι' αυτό το λόγο ζητώ να μην λάβουμε υπόψη μας αυτή την προφορική τροπολογία που εμφανίζεται στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ας ψηφίσουμε απλώς τη συμβαστική τροπολογία 12 χωρίς προφορική τροπολογία και έπειτα η 154 δεν θα καλύπτεται πλέον από τη συμβαστική τροπολογία, άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία αυτή ξεχωριστά ως τροποποίηση ουσιαστικά της προφορικής τροπολογίας. Πρόεδρος. Άρα αν εγκριθεί η 12 θα ψηφίσουμε και την 154. Κατάλαβα σωστά. Πολύ ωραία. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αλλά θα το παληθεύσουμε και ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 154. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. και όντω απορρίπτεται. Ήταν πάντως θετικό το ότι επαληθεύσαμε ηλεκτρονικά. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την ανθρωπολογία 157 άρτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για τροπολογία 169 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Με συγχωρείτε, είναι σε δύο τμήματα αυτή η τροπολογία. Τροπολογία 179 πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 181 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, το πρώτο τμήμα, το πρώτο τμήμα της 182 κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές. Ας την ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 187, άρτη ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 185. Λοιπόν, η 187 εγκρίνεται, 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 189. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 195, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 212, άρχεται ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. 213 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 214 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 214. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υπεράριθμη από το ΕΛΚ. Ένας επιπλέον. Δεν είναι εδώ η Αγγέλ Κανίμπλερ. Τώρα είναι εντάξει. Πέρας λοιπόν απορρίπτεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 222. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Πάλι ένα επιπλέον μέλος από το ΕΛΚ. Πέρας. Εγκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στην ελέγξουμε και ηλεκτρονικά άρτη ψηφοφορία για τη 223. Πέρας. Όντως εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 37 λέει ο υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 37. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 43, άρχιτη ψηφοφορία. Τη 43 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 46 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 47 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 48. Άρχιτη ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 1 υπέρ, κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 1, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 1, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται.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 για τροπολογία 11 από την Επιτροπή Απασχόλησης. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση και για την 18 από την Επιτροπή Απασχόληση. Λυπάμαι, αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια σα καλά, λέει ο Πρόεδρο. Η ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την 18 τη Επιτροπή Απασχόληση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 23 Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο μαζί, 26-27 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. 9 από την Επιτροπή Αλίας ε, υπέρ. Κατά, η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 9 της Επιτροπής Αλίας, άρτη ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται, 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά ηλεκτρονική υπαλλήθευση για τροπολογία 43 της Επιτροπής Αλίας άρτη ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική τώρα ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Συγχαρητήρια στον εισαγητή μας κύριο Φερέιρα. 49 υπέρ, 8 ψήφοι κατά, ουδεμία αποχή. Συγχαρητήρια αγαπητές συνάδελφοι. Interoperability solution. Τώρα λοιπόν πάμε στην επόμενη, ε, στο σημείο υπαριθμών 6, στην ψηφοφορία στις λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες δίκες κτλ. Ο κύριος ε, Ζωρίνιο είναι συγκητή. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΙΜΚΟ 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έλεγχος, ηλεκτρονική επανλήψη. Έκλειση ψηφοφορία. Αποδεκτή. 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 ΙΜΚΟ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 75 υπέρ κατά αποχές ε, κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 75 παρακαλώ. Περισσεύει ένα από το ΕΛΚ παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Αποδεκτή η τροπολογία. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΝΚΟ 36 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ινκο 36 παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η σημαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 14 σημαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η ΙΜΚΟ 39 υπέρ κατάποχες εγκρίνεται. Συμμεστική 16 υπέρ κατάποχες εγκρίνεται. Η 17 υπέρ κατάποχες εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 40 ήταν αυτή. Τώρα η 88 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 93 υπέρ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 1-2-5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1-2-6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. 1-2-6 ψηφίζουμε για την 1-2-6. 1-2-6 παρακαλώ. Έκλεισε η ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. Η 22 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή η 133 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 133 έκλεισε ψηφοφορία απορρίπτεται ΥΜΚΟ 50 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή η 51 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Η 52 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Τροπολογία 134 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 53 ίνκο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 54 ίνκο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 137 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 137. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 138 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση και πάλι παρακαλώ. 138. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έγκληση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ήμκο 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 3 κατά αποχές εγκρίνεται, η 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΜΚΟ 3 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση η ΜΚΟ 3. Πρέπει να ελέγξουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. ΜΚΟ 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΙΜΚΟ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΙΜΚΟ 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 4, 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 45 παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Η 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 47 υπέρ, κατά, Η 47 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκλεισε η ψυχοπορία. Η 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 49. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Για το σύνολο της έκθεσης παρακαλώ ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. 52 υπέρ, 2 κατά, συνάδελφε Ζωρίνιο, συγχαρητήρια για την έκθεσή σας. Και τώρα πάμε στην τελευταία εξίσου σημαντική ψηφοφορία Προεπολογισμό 2016, εντολή για τον τριμερή διάλογο. Ε, συντάκτρια Ανελίν Βαν Μπόσουτ. Λυπάμαι αν την πρόφερα σωστά το όνομά σα. Ξεκινάμε λοιπόν. Συμβεβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε την 9 παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Αφού λέει ο γραμματέας θα το ελέγξουμε. Συμβαστική 9. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά Ελέγχουμε τη 48, άρχεται η ψηφοφορία. Well, Christian, we should be sure about Christian, πρέπει να είμαστε βέβαιοι για το ότι θα γίνει με την τροπολογία σας. Πέρας ψηφοφορίας. Βλέπετε. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο της έκθεσης τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Πολύ καλό το αποτέλεσμα. 46 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 6 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Ανλίν Βαν Μπόσιτ. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Λυπούμε, αλλά τελείωσαν οι ψηφοφορίε. Καλό ή κακό νέο δεν ξέρω. Εξαιρετικό, ε. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Προτεραιότητες τη ήτρε στον προπολογισμό του 2016 ανταλλαγή απόψεων με τον Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε, Γενικό Εισηγητή για τον προπολογισμό του 2016. Συνάδελφο από την Επιτροπή Προπολογισμού.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 Λυπάμαι αγαπητοί συνάλφοι που φεύγετε, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σας σταματήσουμε. And we are also very lucky that colleague, colleague rapporteur is not with us. Co colleague, he's, he's waiting, yes? Okay, good.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 Dear friend Miriam. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητή Μίριαμ, σας παρακαλώ να καθίσετε. Και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που δεν έχουν ακόμη καθίσει, να καθίσουν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σας υπενθυμίζω λοιπόν, το σημείο 8 συζητούμε, προτεραιότητες τη ΣΥΤΡΑ στον προπολογισμό του 2016, ανταλλαγή απόψεων με τον Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε, Γενικό Εισηγητή για τον προπολογισμό του 2016. Καλώ ήλθατε στην Επιτροπή είτε αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι βέβαια στην παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω όμω ότι σε ό,τι αφορά την ε, θέση μας σε ό,τι αφορά ε, τις διαπραγματεύσεις όπως το διαλόγου ψηφίστηκε σήμερα. Η συγκήτρια είναι εδώ στην αίθουσα. Είναι πολύ σημαντικός ο προπολογισμό. αν θέλουμε να έχουν αισιοπέραση οι προτεραιότητες μας που είναι ανταγωνιστικότητα βέβαια της οικονομίας, βιομηχανία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία, ICT, τεχνολογία πληροφοριών, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνίες, δέσμη μέτρων και φυσικά και η ενέργεια. Άρα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν προϋπολογισμό που θα μας επιτρέψει επίσης να έχουμε και μια στρατηγική εξόδου από την κρίση. Πολύ σημαντικό και αυτό σύν την ανταγωνιστικότητα. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 30 με 40 λεπτά για την ε, ανταλλαγή απόψεων αυτή. Θα παρακαλέσω τον συνάδελφό μας, Φερνάντες, εισηγητή, να μας παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2016. Παρακαλώ. Okay, Euh, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γαλλικά. Οι γενικέ κατευθύνσει εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια για τον προπολογισμό του 2016 στις 11 Μαρτίου του 2015. Σας υπενθυμίζω τα τρία «Ε», «Emploi Entreprise» και «Δήμικρο και «Entrepreneurship» απασχόληση, επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα. Αυτές είναι τρεις προτεραιότητες λοιπόν. Ένα α είναι η κύρια κατηγορία. Ε, έχουμε επίσης και την εσωτερική αλληλεγγύη και την πολιτική συνοχής που είναι σημαντική για την εσωτερική αλληλεγγύη. Αλλά και εξίσου σημαντική είναι για την έρευνα, για την ανάπτυξη πολιτική συνοχής και για την απασχόληση. Και εξωτερική αλληλεγγύη βέβαια είναι θέμα. Δεν μπορούμε να λησμονούμε τι συμβαίνει έξω από την Ευρώπη. Και η ασφάλεια, μετανάστευση, επίσης σημαντικές ανησυχίες. Ακινούμε από την εξή αρχή. Το Συμβούλιο ή Κομισιόν θα πρέπει να, δεσ... να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους. Αυτό τι σημαίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να σεβαστούν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως το Συμβούλιο ολισμονεί συχνά ότι έχουμε ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο έχουμε επιτύχει την ευελιξία. Για παράδειγμα, καταφέραμε να έχουμε ένα συνολικό περιθώριο για τις ε, ανεκμετάλλευτες πιστώσεις της προηγούμενης χρονιάς. Είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε πολλές φορές. Το Συμβούλιο δεν ήθελε να χρησιμοποιηθεί αυτό το περιθώριο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Όμως το πετύχαμε και πρόκειται για ένα νεοτερισμό στο πολιετές νοσιονομικό πλαίσιο. Το άρθρο 14, τα ε, περιθώρια ενός έτσι που δεν έχουν ε, χρησιμοποιηθεί, εντάσσονται σε ένα γενικό περιθώριο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολιτικούς στόχους και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θέλουμε λοιπόν αυτή την ευελιξία να τη χρησιμοποιήσουμε, να την αξιοποιήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο εγκρίναμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο παρότι μειωμένο. Γιατί θέλαμε να υπάρχει αυτή η ευελιξία και την διεκδίκηση αυτή την πετύχαμε. Υπάρχουν και όλα τα άλλα μέσα ευέλιξίας βέβαια, που και αυτά είναι σημαντικά, όμως ε, ο σεβασμός των δεσμεύσεων σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσουμε αυτά που πρέπει να πληρώσουμε, γιατί είναι κάπως γελίο να λέμε ότι η αναλήψη υποχρεώσεων, οι δεσμεύσει, όπως είναι και ξεκάθαρο, μεταφράζονται σε πληρωμές. Μα είναι λογικό και επόμενο. Έχουμε ένα σχέδιο πληρωμών, για να μειώσουμε αυτά τα καθυστερούμενα στους ανεξόφτους λογαριασμούς, συμφωνήσαμε για το 2016 να μην έχουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ανεξόφλητους λογαριασμούς στο πλαίσιο 2006-2013. Το προηγούμενο δηλαδή δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης συμφωνήσαμε για το ΕΦΣΙ να μειωθεί ο αντίκτυπος στο Connecting Europe και στο ορίζοντα 2020 ένα δις αντί για έξι δις είναι οι περικοπές. Πέντε δις μόνο. 23 Ιουνίου, να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα, εγκρίνουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών την έκθεση, η εντολή για τον τριμερή διάλογο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια 3 Σεπτεμβρίου για την κατάθεση τροπολίδων μέσα Σεπτεμβρίου. Οι γνωμοδοτήσεις για το ψήσιμο του Οκτωβρίου 28-29-30 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε στην Επιτροπή Προπολογισμού. 12-13 Οκτωβρίου ψηφίζουμε το ψήφισμα 28 Οκτωβρίου στο ψηφίσμα στην επιτροπη προπολογισμου 12 13 οκτωβριου ψηφιζουμε το ψησιμο 28 οκτωβριου στο ψηφισμα στην ολομελεια Και τον Νοέμβριο η συνδιαλλαγή. Πολύ γρήγορα σε ό,τι το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πευλήθησης στις 27 Μαΐου. Το Συμβούλιο βέβαια ξέρετε ότι πρέπει να προβεί στην ανάγνωση του σχεδίου προπολογισμού και να τοποθετηθεί ό,τι αφορά την Επιτροπή σας για το κόσμο. 4,8% μειώθηκε ε, το ποσοστό των αναλήψεων υποχρεώσεων σε σχέση με το 2015 για τον ορίζοντα 2020. 1,9 είναι η ανέλυψη να θα αλλάξει αυτό γιατί στην τελική συμφωνία μειώθηκε αυτό προς τον περικοπών για τον ορίζοντα 2020. Σε πληρωμές όμως έχουμε αύξηση τάξη στο 11,6% για τον ορίζοντα 2020, άρα ένα δις. Οι πληρωμή είναι σημαντικό ζήτημα. Θέλουμε να έχουμε επαρκή κονδύλια για τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Έρχομαι στους οργανισμούς. Αυξήθηκαν τα ποσά. Όπως και τα προηγούμενα χρονιά είχαμε ε, καταλήξει ένα συμβιβασμό και για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουμε ένα περιθώριο στο 1α που μειώθηκε και με τη συμφωνία για το ΕΦΣΥ, γιατί τα περιθώρια τα χρησιμοποίησαμε για να μειωθεί ο αντίκτυπος στον ορίζοντα 2020. Βέβαια τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν ένα άλλο όριο, 140 εκατομμύρια για όλες τις προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά προγράμματα, 100 εκατομμύρια για τις προπαρασκευαστικές ανάγκες και 40 εκατομμύρια για τα πιλωτικά προγράμματα. Συνολικά, μπορώ να πω ότι είναι κακό το αποτέλεσμα, πρόκειται όμως για ένα συμβιβασμό. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας και τι σημαίνει αυτό, ότι σε κάθε δημοσιονομική διαδικασία, σε κάθε διαδικασία ε, κατάθεσης του υπερπολισμού κάθε χρονιά θα προσπαθούμε να μειώνουμε όσο θα δούμε περισσότερο τον αντίκτυπο ε, στη διευκόλυνση Connecting Europe, σύμφωνα στην Ευρώπη, και στον ορίζοντα 2020. Θέλουμε να έχουμε βέβαια το Ταμείο και θέλουμε και τη δική σας υποστήριξη και την δική σας δέσμευση ως Επιτροπή για να δούμε ποιες είναι οι θέσεις που πρέπει και τα κονδύλια που πρέπει να περασπιζόμαστε κάθε χρόνο. Και επαναλαμβάνω κυρίως για τον ορίζοντα 2020, διότι καταφέραμε να έχουμε συν ένα δισεκατομμύριο για αυτά τα προγράμματα. Αλλά δεν έχει τελειώσει το πράγμα, διότι από την αρχή είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και το Συμβούλιο, πολλές φορές ξεχνάνε ότι την προκοδότηση του Ταμείου την κάνουμε ε, κάθε χρονιά και υπάρχει και η δημοσιονομική ευελιξία που περιλαμβάνεται στη διοργανική σύμφωνη. Μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε οι δύο αρχές επί του προπολογισμού ένα πρόγραμμα, μπορούμε να το μειώσουμε να το αυξήσουμε κατά 10%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η δική μας δουλειά και η δική μας μάχη θα συνεχιστεί στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Uh, thank you. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Να ζητήσω τώρα από, τον, από τριά μας, την κυρία Νελίν Βαν Βοσούτ, να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Φερνάντε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι όντω ε, η συγγήτρια για την Επιτροπή Βιομηχανία όσον αφορά τον προπολογισμό 2016 και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το ότι βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια σημαντική συνένεση όσον αφορά τις προτεραιότητες τις προτεραιότητες δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έτος 2016. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη και τη γνωμοδότησή μας, αυτή την οποία εγκρίναμε μόλις πριν από λίγο με 48 ψήφους υπέρ και δύο μόνο κατά. Φαίνεται λοιπόν ότι η Επιτροπή Βιομηχανίας στηρίζει σχεδόν ομόφωνα τις προτεραιότητες που έχουμε εμείς για το 2016. Ορίζοντας 2020 είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία περικοπή ούτε καν για τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Ξέρετε ότι εδώ και δύο χρόνια διαπραγματευόμαστε σκληρά για το πρόγραμμα αυτό και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Προγράμματα όπως ορίζοντας 2020 το ΣΕΦ, η διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, ιδίως την έχουν απαιτήσει Τόσε πολλέ διαπραγματεύσει και όταν επιφέρουν τέτοια σημαντική προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη δεν θα, πρέπει να περικόπτονται κατά αυτόν τον τρόπο και τόσο δραστικά. Πολύ φοβάμαι ότι όταν κάνουμε κάτι τέτοιο στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν εμεί ω Επιτροπή Βιομηχανία μια καλύτερη ρύθμιση όσον αφορά τα προγράμματα αυτά και νομίζουμε ότι για την προσέγγιση αυτή δεσμεύεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία από ό,τι φαίνεται θέλει να διατηρήσει αυτά τα δύο προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσει να δεσμεύεται πλήρω τόσο για τον ορίζοντα 2020 όσο και για τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν εμείς να μας βεβαιώσετε ότι κι εσείς αυτήν ακριβώς τη θέση θα υποστηρίξετε ως εισηγητής για το 2016. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει προταθεί, τι θα προταθεί στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου για τα δύο αυτά προγράμματα, αλλά θα θέλαμε τη διαβεβαίωση ότι εσείς είστε με το μέρος μας, ότι ασπάζεστε τη δική μας την άποψη. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ενεργειακή αποδοτικότητα, τα μέσα διασύνδεσης, η ενεργειακή ένωση, η εξοικονόμηση ενέργειας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των ανεξόφλητων λογαριασμών και της καθυστέρησης στην καταβολή των πληρωμών. Ποιες λοιπόν οι προτεραιότητες για το 1α του προπολογισμού και τι θα κάνετε με τις δικές μας τις προτεραιότητες. Θεωρείτε ότι συνάδουν με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Προπολογισμών. Και ένα ακόμα ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει η δική μας Επιτροπή προκειμένου να υποστηρίξει τις δικές σας αρχές. Ξέρω ότι ε, μέχρι τις 18 Αυγούστου μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες όσον αφορά τις γραμμές του προπολογισμού που θέλετε εσείς να προασπίσετε. Μπορείτε να μας πείτε εσείς τι είδους τροπολογίες θα θέλετε από τη δική μας την Επιτροπή, τι θα σας διευκόλυνε εσάς το έργο που πρέπει να επιτελέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Οι σκιώδεις ηγητές έχουν το λόγο. Κάριτς, μάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο δικός μας ο σκιοδησηγητής δεν είναι εδώ, απλά θέλω να επαναλάβω ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να πω ότι μόλις ψηφίσαμε στην Επιτροπή μας για όλα τα θέματα ε, τα οποία είναι επίμαχα στις ε, πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά αυτό δεν είναι ένα από αυτά. Κατά την τελευταία θητεία ε, κατεβλήθησαν πολύ μεγάλες ε, προσπάθειες για να επιληθούν τα προβλήματα. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Αν σας κατάλαβα καλά, είπατε ότι στον προεπλογισμό του 2016 είναι ότι θα υπάρχει ένα έλλειμμα, δηλαδή μια διαφορά ανάμεσα στις πλωμές και τις υποχρώσεις του μεγέθους των 2 δις ευρώ. Αυτό όμω ε, ανησυχεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι δηλαδή ε, ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακριβώ αυτό το κενό ανάμεσα στι υποχρώσει μα και τι πληρωμέ. Και θεωρώ ότι μπορούν να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και αυτό θα βοηθήσει όλα τα προγράμματα και σίγουρα και το Horizon 2020. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών, η κυρία Μούντι. Ε, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Σας βλέπουμε ε, σε ταυτόχρονα κατευθύνματα στην Επιτροπή Προβλητισμών, αλλά όχι εδώ. Καλωσορίσατε λοιπόν. Όπως ε, γνωρίζετε, υπάρχει ευρία συνένεση για το πού ακριβώς θέλουμε να κατευθυνθούμε με τον προϋπολογισμό του 2016. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το να βλέπει κανείς πώς οι πολιτικές ομάδες και οι διάφορες επιτροπές συνεργάζονται προσπαθούν ε, να προστατεύσουν το πρόγραμμα 2020. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μέσω των ε, διαπραγματεύσεων και να διασφαλίσουμε ότι στο πρόγραμμα Horizon 2020 θα αναγνωρίσουμε και θα στηρίξουμε τη, το, τη διαφορά αυτή που υπάρχει και αφορά τόσο στις επιδοτήσεις όσο και στα οικονομικά εργαλεία όπως είναι το ε, Ταμείο Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Η τα κονδύλια για επιδοτήσεις ε, δεν αφορούν μόνο το πρόγραμμα Marie Curie, αλλά και άλλα προγράμματα, άλλους τομείς ε, του ε, προγράμματος Horizon 2020. Άρα δηλαδή, επειδή όπως πολύ συχνά ε, λέμε ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες και καθώς πλησιάζουμε τις ε, τελικές διαπραγματεύσεις αυτό επαληθεύεται όλο και περισσότερο. Ε, θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε γενικά για το Horizon 2020 αλλά και όσον αφορά τις διαφορές, τις μικρές λεπτομέρειες που αφορούν στο πρόγραμμα Horizon 2020. Ε, Ο συνάδελφος Γκαλμπράντε από την Άλντα, από τις Φιλελεύθερες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σε ευχαριστούμε κύριε Φερνάνδες που ήρθατε και η δική μου η ερώτηση έχει σχέση με το πρόβλημα των πληρωμών. Το είπατε και εσείς ο ίδιος ε, και το ρώτησαν και άλλοι συνάδελφοι και θέλω να σας ερωτήσω πολύ συγκεκριμένα σχετικά με το πρόγραμμα πληρωμών το οποίο έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν είμαι σωστά ενημερωμένος, η Κομισιόν βάζει προτεραιότητες στις πληρωμές ε, όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και στις καινοτομίες ε, και, τις, και στην έρευνα και εκεί υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς αυτό το αναγνωρίζετε και πιστεύετε όπως και εγώ ότι η δυνατότητα απορρόφησης ε, των κρατών μελών στο πλαίσιο της ε, ε, πολιτικής συνοχής είναι ένα πρόβλημα και οι πληρωμές, τα κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία είναι διαφορετικού μεγέθους και διαφορετική σημασία. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει εδώ να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τώρα τους υπόλοιπους ομιλητές, αλλά και η κυρία Βαν Μπρέντ είναι η συγγήτρια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο βέβαια είναι, όπως γνωρίζετε, πάρα πολύ σημαντικό. Τη δίνω λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το ΕΦΣΥ στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Ξέρετε ότι είναι τεράστιος ο αντίκτυπος στον ε, προπολογισμό. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Φερνάντες για τη μάχη που δώσαμε από κοινού κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων. Δώσαμε την ίδια μάχη θεωρώ και ήταν πολύ σκληρή η μάχη αυτή. Μολονότι είχαμε μια σημαντική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο με τους συναδέλφους από την Ήτρε, την Τραν και από την Επιτροπή Προπολογισμών, καθώς επίσης και με συναδέλφους από άλλες επιτροπές, είχαμε δημιουργήσει ένα τείχος για να προασπίσουμε όλα αυτά τα οποία θεωρούμε ότι έπρεπε να προασπίσουμε στα πλαίσια του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη και του ορίζοντα 2020. Και είχαμε έπειτα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο διαδραμάτισαν το ρόλο που διαδραμάτισαν κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων και μου προκάλεσε έκπληξη και θέλησα και απογοήτευση το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θέλησαν να αναλάβουν κάποιε δεσμεύσει όσον αφορά τι δραστηριότητε έρευνα και όσον αφορά τα προγράμματα τα οποία υπάγονται στον ορίζοντα 2020 και μάλιστα έδειξαν και πολύ μειωμένη γνώση όσον αφορά τα προγράμματα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι καταφέραμε να περισσώσουμε ό,τι μπορούσε τελικά να σωθεί. Το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι ποσό το οποίο θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε. Πάντως στα πλαίσια των μελλοντικών διαπραγματεύσεων, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρώτον, υπάρχουν δύο μηνύματα τα οποία θα ήθελα να στείλω προς εσάς αλλά και προς υπόλοιπους συναδέλφους. Πρώτον, υπάρχει ακόμα μια διάσπαση όσον αφορά τον ορίζοντα 2020. Από τότε που εμείς διατηρήσαμε μια πολύ ισχυρή στάση λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε ποια μορφή θα πρέπει να πάρει το πρόγραμμα αυτό. Ο προπολογισμό 2016 και όλε οι σχετικέ ομάδε εργασία θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει επιτέλου ποιε είναι οι δικέ μα προτεραιότητε. Και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η κυρία Γεωργίευα, η Επίτροπο, μου είπε ατύπως ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα περιθώριο ευελιξίας όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 και την κατάτμιση ε, κονδυλίων που προβλέπεται εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε έπειτα τι θα γίνει όμως με τον προπολογισμό του 2016 και για την περίοδο μετά το 2016. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να αποδεχθώ τις περαιτέρω περικοπές που προβλέπονται και ότι έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία και θα πρέπει να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα θα πρότεινα να εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνουμε ένα μάχη, αν μη τι άλλο σε αιτήσια βάση, προκειμένου κάθε χρόνο να έχουμε επιστροφή κονδυλίων στον ορίζοντα 2020 και στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτό το μήνυμα νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε και προς τους συναδέλφους της Επιτροπής Προπολογισμών. Δεν είμαι ειδική σε θέματα προπολογισμού, αλλά στα πλαίσια διαπραγματεύσεων συνειδητοποίησα ότι ως Επιτροπή Ήτρα ακριβώς αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Να ακολουθήσουμε δηλαδή τη συμβουλή που μας δώσαν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Προπολογισμών και να απαιτούμε επιστροφή κονδυλίων στα προγράμματα αυτά κάθε χρόνο. Ο κύριος Φέντερ έχει το λόγο σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω και εγώ ότι πραγματικά η Επιτροπή μας στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουμε τα επόμενα χρόνια όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και όσον αφορά και τον ορίζοντα 2020. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί παράλληλα δύο πρωτοβουλίε. Πρέπει να δούμε πώ θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε τι πρωτοβουλίε αυτέ, συμπεριλαμβάνοντα και την πρωτοβουλία για την Ενεργειακή Ένωση. Νομίζω ότι στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για το ΕΦΣΥ στείλαμε και εμείς ως Επιτροπή Ήτρε ένα πολύ χειρό μήνυμα και είπαμε όπως και συνάδελφοι από άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές ότι μολονότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποια περιθώρια από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν θέλουμε να γίνουν περικοπές από τον ορίζοντα 2020 γιατί είναι το μόνο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τις εργασίες του αύριο και οποιαδήποτε προοπτική οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να παρατείνουμε την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να εστιαζόμαστε όλο και περισσότερο στο μέλλον και νομίζω ότι η έρευνα και η κοινοτομία βρίσκονται στην καρδιά οποιασδήποτε μελλοντική προπτικής για ανάκαμψη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιο άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που ήλθατε κύριε Φερνάντες Χθε στην ΕΚΟ στην ίδια συζήτηση θα θέλαμε να είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρούσα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορα σημεία. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε δηλαδή για πολλά σημεία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του προπολογισμού, όπως για παράδειγμα ότι η δική μας ομάδα δεν συμφωνεί με το σχέδιο Juncker και ιδίω με το πώς τελικά προωθούμε την ε, κερδοσκοπική ανάπτυξη, αν μπορώ να το πω. Δεν θέλω να μιλήσω για τον περιπολισμό γέννη, να, να περιστώ ε, στο κόσμο. Μιλάμε για περικοπές εδώ και είναι απαράδεκτο το μόνο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που στόχο έχει τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ που είναι πάνω από το 60% του επιχειρηματικού ιστού να έχει περικοπές. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να ορίσουμε μια συμπεριφορά και μια στάση για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αλληλέγγυο ώστε οι ανεξάρτητοι συνεταιρισμοί που δεν είναι οι μεγάλες πολυεθνικές να μπορούν τις δραστηριότητες τους να τις προσανατολίζουν για, το κοινό όφελο, το όφελο της κοινωνίας και σε συνεργασία με το δημόσιο τομέα. Σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία χαιρόμαστε που υπάρχει αύξηση των κονδυλίων, όμως σε ό,τι αφορά τους όρους εφαρμογής των προγραμμάτων δεν συμφωνούμε που δίνεται προτεραιότητα στην πρόσβαση σε πίστη, ε, σε δάνες, αυτούς που δεν το χρειάζονται ουσιαστικά, δηλαδή στις μεγάλες πολυεθνικές από το μισό από η φαρμακοβιομηχανία, πως αυτά τα προγράμματα βρίσκουν μια νέα κερδοφόρα αποκλειστική αγορά και δεν προωθούμε το συνεταιρισμού ε, ή τι μικρές ε, επιχείρησεις στους μικρούς ερευνητές. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει την έρευνα να την ε, βάλουμε να υπηρετεί μια μερκαντιλιστική λογική. Αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε το κοινωνικό της έργο. Ευχαριστώ. Oh, Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς άλλο το λόγο. Επομένως, κύριε Φερνάντες, μπορείτε να πάρετε το λόγο για να συνοψίσετε λίγο τη συζήτηση αυτή και να καταλήξετε σε κάποια συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά για την συμβολή σας στη συζήτηση αυτή. Δεν είμαι εγώ που θα πω βέβαια στην Επιτροπή Βιομηχανίας ποιες τροπολογίες πρέπει να υποβάλει ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν μπορώ να δώσω τέτοιες υποδείξεις εγώ στους συναδέλφους μου. Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ποιες τροπολογίες ε, οφείλετε να υποβάλλετε. Άκουσα πάντω ποιε ήταν οι σα, σας. Ξέρω ότι το τμήμα 1α του προπολογισμού αποτελεί για εσά πολύ σημαντική προτεραιότητα τόσο για το στόχο τη απασχόληση όσο και για το στόχο τη υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και για το στόχο τη λεγόμενη επιχειρηματικότητα, του επιχειρηματικού αυτού πνεύματο που πρέπει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ πάντω θα παρακολουθήσω πολύ στενά όλες τις εξελίξεις προκειμένου να καταφέρουμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους στόχους που νομίζω ότι μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Όλοι συμφωνούμε με αυτά τα τρία ε. Όσον αφορά τώρα τον ορίζοντα 2020, στην αρχή των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να θυμηθείτε ότι ουδείς, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο, θέλουν να αλλάξουν το παραμικρό. Τίποτα απολύτως δεν θέλουν να αλλάξουν όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Το να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δισεκατομμύριο ευρώ, να καταφέρουμε δηλαδή να περισσώσουμε το ποσό αυτό, ήταν στην αρχή ένας απίστευτος άθλος που δεν πιστεύουμε ότι θα καταφέρναμε να πετύχουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν τη συμβολή της συναδέλφου Βαν Μπρέντ γι' αυτό και καταφέραμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα μη χρησιμοποιημένα περιθώρια από το γενικό περιθώριο, το οποίο δεν ήθελε καν να αναφέρει, δεν ήθελε καν να θίξουμε το Συμβούλιο. Είχαμε πάντως δίκιο που επιμείναμε και αξίζει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό και στο μέλλον. Επίσης, στον κανονισμό της δημοσιονομικής διαδικασίας κάθε φορά είπαμε ότι θα πρέπει να βλέπουμε τι μπορεί να γίνει με τη χρηματοδότηση του Ταμείου. Και αυτό αρχικά δεν το ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο. Και Όσον αφορά έπειτα το άρθρο εκείνο που έχει να κάνει με την επιλογή των συγκεκριμένων σχεδίων, ε, νομίζω ότι ήταν το άρθρο 5.2, αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει κάπως η ρύθμιση, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο υφιστάμενος τώρα αριθμό, πάντως αναφέρομαι στις προτεραιότητες εκείνες ε, της έρευνας, τις οποίες έχετε υποστηρίξει και εσείς ως Ήτρε. Καταφέραμε λοιπόν να προασπίσουμε τις προτεραιότητές σας και στα πλαίσια του κανονισμού. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί τον κανονισμό θα χρησιμοποιήσουμε και για τον τομέα της έρευνας. Και κάτι ακόμα. Καταφέραμε να προστατεύσουμε τις γραμμές προπολογισμού για τη βασική θεμελιώδη έρευνα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα ήμουν καθόλου σοβαρό αν σας έλεγα ότι τα 2-7 δισεκατομμύρια ευρώ μπορούμε να τα έχουμε από τη μία μέρα στην άλλη και στα πλαίσια της υφιστάμενης δημοσιονομικής διαδικασίας, δηλαδή μέχρι το 2016. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι γραμμές του προπολογισμού που θα πρέπει να προασπίσουμε στα πλαίσια της τρέχουσας και της μελλοντικής δημοσιονομικής διαδικασίας, προκειμένου να καταφέρουμε να μειώσουμε οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση που θα έχουν οι μελλοντικοί προπολογισμοί στον τομέα της έρευνας. Νομίζω ότι Εκεί ακριβώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτέ τι συγκεκριμένε γραμμέ προπολογισμού και σε σχετικά ποσά. Α ξεκινήσουμε ήδη από το 2016. Σίγουρα ο δρόμο θα είναι μακρύ και γι' αυτό το λόγο χρειάζομαι και τη δική σα τη δέσμευση, τη δική σα την υποστήριξη, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και είμαι σίγουρος ότι ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική συνένεση. Δεν ξέρω βέβαια θα καταφέρουμε να πετύχουμε και τη συνένεση αυτή όσον αφορά τη γραμμή του προπολογισμού που θα πρέπει να προστατεύσουμε. Δεν μπορώ όμως εγώ να υποδείξω ποια θα είναι αυτή η γραμμή του προπολογισμού. Εναπόκειται σε εσά να καταλήξετε σε μια συμφωνία για τίνη τις γραμμές προπολογισμού και τα σχετικά ποσά που θα πρέπει να προασπίσουμε στα πλαίσια του προπολογισμού 2016 και των μελλοντικών προπολογισμών. Πάντω, στόχο μα σε κάθε περίπτωση είναι να μειώσουμε οποιαδήποτε οικονομική επίπτωση για τον ορίζοντα 2020 και το μέσο συνδέοντα την Ευρώπη. Και είναι τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ήταν το μόνο που υπεράσπισε τα δύο αυτά προγράμματα, τα οποία τη χάνουν διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια στιγμή πραγματικά είχα αποθαρρυνθεί και νόμιζα ότι θα καταφέρναμε να εξασφαλίσουμε αυτό το δισεκατομμύριο ευρώ. Το πετύχαμε όμω. Όσον αφορά τι πληρωμέ, δεν υπάρχουν προτεραιότητε για τι πιστώσει πληρωμών. Έχουμε προτεραιότητε για τι πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων. Οι πληρωμέ αποτελούν λογικό επακόλουθο των δεσμεύσεών μα, των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε. Όσον αφορά τώρα την πολιτική συνοχή, ε, τομέα 1β, ξέρετε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ σημαντική καθυστέρηση στι πληρωμέ και στην εξόφληση των λογαριασμών. Είναι λοιπόν λογικό να δώσουμε εκεί περισσότερα χρήματα προκειμένου να θεραπεύσουμε το πρόβλημα αυτό και να καταφέρουμε να καλύψουμε αυτό το υψηλότατο ποσό καθυστερημένων πληρωμών στον τομέα 1β θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί είναι οι κανόνες. Αυτά επιβάλλει ο κανονισμός και ο κανονισμός του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που λέει ότι στα πλαίσια των πληρωμών για την πολιτική συνοχή έχουμε τον κανόνα 1 συν 3. Αυτός είναι ο κανόνας που ισχύει και αυτός είναι ο κανόνας τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Ας μην το ξεχνάμε, αυτό ισχύει από όλο το κανόνας αυτός 1 συν 3 για την πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή σε πάρα πολλέ χώρες, ας μην το ξεχνάμε αυτό, συμβάλλει και στην ίδια την έρευνα. Η πολιτική συνοχή συμβάλλει και στην ευφυή ανάπτυξη. Δεν έχουμε μόνο απλώς κάποιες επενδύσεις. Αν δούμε το λειτουργικό πρόγραμμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την πολιτική συνοχή σε διάφορες χώρες, θα συνειδητοποιήσουμε ότι τα περισσότερα κονδύλια πηγαίνουν στην οικονομική ανάπτυξη, πηγαίνουν στην απασχόληση, υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ίδια την έρευνα. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τη μάχη αυτή για να διασώσουμε τα κονδύλια του ορίζοντα 2020 καθώς επίσης και τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε τη μάχη αυτή και είμαι σίγουρο ότι θα έχω και τη δική σας την στήριξη. Τώρα για το πρόγραμμα COSME. Εδώ υπάρχει όντως μία μείωση, μία περικοπή στα κονδύλια, το αποδέχομαι κι εγώ, αλλά επισήμως δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, γιατί είχαμε μία προκαταβολή κάποιων ποσών. Και ακριβώ επειδή υπήρξε αυτή η προκαταβολή ποσών, δημιουργεί η εντύπωση τα επόμενα χρόνια ότι έχουμε λιγότερα κονδύλια. Αν πάρουμε όμως ε, το σύνολο των κονδυλίων υπόψη μας, θα δούμε ότι δεν υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά. Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει κατά προτεραιότητα να υποστηρίξουμε και αυτό το πρόγραμμα οι δικέ μου προτεραιότητε, τι οποίε βλέπετε στην έκθεσή μου όσον αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο, νομίζω και δικέ σα προτεραιότητε, αλλά προφανώ θα λάβω υπόψη μου και τη γνωμοδότησή σα. η οποία θα ενσωματωθεί σε αυτό το σχέδιο έκθεση το δικό μου, το οποίο θα ψηφιστεί, όπως σας είπα, την επόμενη εβδομάδα στις 23 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χωσέ Μανουέλ, αγαπητέ συνάδελφε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν τόσο συγκεκριμένο στι προτεραιότητε αυτέ που μας παρουσίασε για τον προπολογισμό του 2016. Όλη αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική για μα και δίνουμε κι εμείς μια μάχη προκειμένου να προωθήσουμε μια στρατηγική εξόδου από την οικονομική κρίση. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα και σου εύχομαι κάθε επιτυχία στην Επιτροπή Προπολογισμών and for great cooperation. Thank you. Uh, um, συνάδελφοι, να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της διάταξη πριν βέβαια από το μεσημεριανό διάλειμμα. Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι. Σον Κέλλιν είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης. Υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής η ΕΝΒΗ και της Επιτροπής ΙΤΡΕ. Διότι έχουμε κοινέ αρμοδιότητες, αλλά υπάρχουν και κάποιες αποκλειστικές αρμοδιότητες. Σε εμά, για παράδειγμα, είναι η έρευνα, η διαρροή άνθρακα, η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η βιομηχανία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όπως είπα έχουμε και κοινέ αρμοδιότητες με την Επιτροπή ΕΜΒΗ. Έχουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα βασίζεται σε έκθεση ίδιας πρωτοβουλία ε, της Επιτροπής ΕΝΒΗ αλλά θα γνωμοδοτήσουμε. Και υπάρχει και προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών και ψηφοφορία στην Επιτροπή μας πολύ στενές προθεσμίες, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν μένουν πολλές εβδομάδες πριν από την παρουσίαση της έκθεσης στην Επιτροπή, άρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ξεκινάει η συζήτηση τώρα, έχουμε 45 λεπτά Αυτός είναι ο χρόνος που προβλέπεται για τη συζήτηση αυτή. Θα παρακαλέσω τον εισηγητή, τον συντάκτη, τον ομοδότη, τον κύριο Σον Κέλλη, να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που είπατε ποια είναι η θέση με μεταξύ επιτροπών ή τρένβη, το, την προθεσμία κατάσταση τροπολών κτλ. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη η σημερινή συζήτηση, ιδίω μετά από τις ε, συζητήσει των τελευταίων ε, εβδομάδων. Πολλές ε, αναφορές λένε ότι δεν υπήρξε ίσως παραπογοητευτική πρόοδος, όμως μπορούμε να αντλήσουμε κάποια ενθάρρυνση από το γεγονός ότι υπήρξε εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις αυτές και είναι σημαντική εμπιστοσύνη. Στο σχέδιο γνωμοδότησης αναφέρω τη σημασία του να έχουμε δεσμευτική παγκόσμια συμφώνια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι η βάση και πρέπει να το πετύχουμε στο Παρίσι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία, την παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία για να πιάσουμε το στόχο των δύο βαθμών Κελσίου. Και θα πρέπει να το δούμε με θετική νοοτροπία, να υπογραμμίσουμε με τι ωφέλη συνεπάγεται αυτό για τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων, νέων θέσεων εργασία, για την ενίσχυση της ε, οικονομικής ανάπτυξης ή δράσεις για την κλιματική αλλαγή συμβαδίζουν με την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να θυμόμαστε επίσης τι σοβαρές επιπτώσεις θα είχε η αδράνεια σε αυτή τη χρονική στιγμή και θα πρέπει και οι ομόλογοι μας από ολόκληρο τον κόσμο να αντιληφθούν το ζήτημα σε, όλη του, ε, σε όλες τις διαστάσεις. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς δεσμεύσεις. Αλλά και οι ανταγωνιστές μας θα πρέπει να δεσμευτούν. Δεν θα πρέπει να είμαστε σε μια θέση όπου τη δική μας φιλοδοξία δεν θα την ακολουθήσουν άλλοι θα πρέπει και άλλες χώρες να γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα χαράς να ηγηθεί ως συνήθως με την προπόθεση όμως ότι θα είμαστε οι μόνοι οι οποίοι θα δράσουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό μέτωπο, σε αυτό το πολύ σημαντικό αγώνα. Και έρχομαι στη διαρροή άνθρακα. Πιστεύω ότι αργότερα θα χρειαστεί να εξασφαλίσουμε ότι θα προβληθούν κάποια μέτρα για τη διαρροή άνθρακα για να καλυφθεί το ενδεχόμενο άλλες χώρες να μην προβούν σε αντίστοιχες δεσμεύσεις. Θα πρέπει να φροντίσουμε ότι οι βασικοί μας τομείς ε, θα τύχουν τις απαραίτητες προστασίας και ότι θα διατηρηθούν θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη, αλλά όχι πολιτικές που θα βλάπτουν το περιβάλλον, επειδή θα υπάρχει ε, μια πιο χαλαρή προσέγγιση σε κάποιους άλλους τομείς ιδίως για τον γεωργοδιατροφικό τομέα είναι σημαντικό αυτό. Θα ήταν αντιπαραγωγικό για τη συλλογική μας δράση στον τομέα της ε, αλλαγής του κλίματος, ιδίως όταν αυξάνεται ο πληθυσμός και χρειάζεται παραγωγή περισσότερων τροφίμων, αλλά και βελτιωμένη απόδοση, να μην ε, καταλήξουμε σε μια δεσμευτική συμφωνία. Η διαρροή του άνθρακα δεν θα έπρεπε να είναι θέμα καν εάν το πετύχουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά το σύστημα εμπορίας ε, δικαιωμάτων εκπομπών, ήταν αποτελεσματικό για τη μείωση του επίπεδου εκπομπών. Βέβαια χρειάζεται ανανέωση αυτό το σύστημα και θα πρέπει να φροντίσουμε ότι αποτελεσματικά πετυχαίνει τους στόχους του. Και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια παγκόσμια αγορά εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Πολύ πρόσφατα το ζήτησε και η ίδια Γερμανίδα καγκελάριος αυτό, η Άγγελα Μέρκελ. Αν έχουμε παντού το ίδιο πλαίσιο θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και στη μείωση εκπομπών και στη βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Θα βελτιωθεί το μέγεθος ε, της αγοράς, θα δοθούν οι απαραίτητοι πόροι και θα διατεθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα Στου τομεί τη αγοράς και τη βιομηχανία. Προφανέ βέβαια είναι ότι θα πρέπει να λειτουργεί σωστά το σύστημα αυτό στην Ευρώπη και μετά να σκεφτούμε την δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος. Πρόσφατα υπήρξαν εκκλήσει και εκφράστηκαν φόβοι για κάποιες επιδοτήσεις οικονομικές που είναι επιλάβεις για το περιβάλλον. Σε πολλές μελέτες έχουμε δει ότι αποτρέπουν τον ανταγωνισμό, αλλά επηρεάζουν και αρνητικά την καινοτομία αυτές οι επιδοτήσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια σταδιακή κατάργησή τους, ιδίως αν θέλουμε να αυξήσουμε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, στο ενεργειακό μείγμα. Πρέπει να υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, ώστε νέες καθαρές τεχνολογίες να μπορέσουν να ευμερίσουν. Καταπολεμήσουμε τις, τις κλιματικές αλλαγές. η καινοτομία στην τεχνολογία. Είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Μπορεί να δώσει και όθηση για τις καθαρές ενέργειες που είναι στόχος και θα βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους για, τις, για την αλλαγή του κλίματος. Θα είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα το να επιμείνουμε στην καινοτομία στις ε, τεχνολογίες αυτές. Ήδη σε πολλές καθαρές τεχνολογίες ενέργειας έχουμε ηγετικό ρόλο. Ο πρόεδρος Γιούνκερ αναφέρε ότι ε, θα πρέπει η Ένωση να είναι παριθμόν ένα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προστατευτούν σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσία και τεχνολογία. Σίγουρα χρειάζεται αυτή η ανταλλαγή, αυτή η μεταφορά τεχνολογία δύο στι αναδυόμενε χώρε. Θα πρέπει να φροντίσουμε όμω ε, κοινοτόμε βιομηχανίε μα να διατηρήσουν πραγματικά δικαιώματα και δικαιώματα δημιουργού. Χαιρετίζουμε επίση το ότι στη συμφωνία αναγνωρίζεται ο σημαντικό ρόλο της βιοενέργειας για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θέλουμε και βιώσιμη παραγωγή βιομάζας και αϊφόρες πρακτικές διαχείρισης των δασών, των δασικών εκτάσεων. Και έχουμε και τα μέτρα για την ε, παγίδευση και αποθήκευση του άνθρακα που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Επίσης χαίρομαι που αναγνωρίζεται σωματικός ε, ρόλος ε, του τομέα της χρήσης γης στην έκθεση του κυρίου Παναγιώ. Τέλος, είναι σημαντικό να δούμε και τα άλλα συμβαλόμενα μέρη τη συμφωνίας. Είπα, Κίνα, δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο της, ώστε αυτά τα θετικά μηνύματα να γίνουν δεσμεύσεις το Δεκέμβρη. Θα πρέπει να είμαστε ισχυροί και να ζητήσουμε να ακολουθήσουν ε, το παράδειγμά μας και να μειώσουν τις εκπομπές τους και οι τα άλλα μέρη. Εμείς μιλάμε για 40% μέχρι το 2030 μείωση. Και μέχρι το 2050 θέλουμε μείωση των εγχώριων εκπομπών κατά 80% σίγουρα Σε επόμενους ε, μήνες όσο χρειαστεί να αναθεωρήσουμε τους στόχους του 2030. Ο εισηγητή Πανιός ζητά αναθεώρηση κάποιων στόχων. Διακόπτεται ο μιλτής. Μα ολοκληρώνω μια πρόταση ακόμη. Νομίζω θα ήταν αντίθετα καλύτερα να παραμείνουμε φιλόδοξοι. Είναι πολύ σημαντικό το μονοπάτι που έχουμε ακολουθήσει και ελπίζω στο Παρίσι να καταλήξουμε συμφωνία. Η κυρία Κέρλτον Ντάρλινγκ εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε από εκεί. Η δουλειά με τους εισηγητές ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό. Επίσης, ε, θέλουμε να αναφέρουμε ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδείξει τον δρόμο όσον αφορά ε, τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή, να υπάρξει δεσμευτική συμφωνία, συμφωνίες με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και παρότι δεν αναφέρεται στο κείμενο υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκηνικό ε, είναι απαραίτητο το σύστημα της ανταλλαγής εκπομπών να βελτιωθεί με στόχο να υπάρχει μια παγκόσμια αγορά. Τώρα, Υπάρχει το θέμα των ε, επιδοτήσεων που παρεμποδίζουν τη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία, κυρίως στους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας. Και ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο του τομέα της βιοενέργειας. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία που θέλουμε και να τα δούμε τα μεν, αλλά κάποια άλλα τα αμφισβητούμε. Πρώτον, παρότι υπάρχει μια αλλαγή ε, ως αποτέλεσμα των συζητήσεων των συντονιστών υπάρχει μια θετική προοπτική στο σχέδιο της ε, γνωμοδότησης. Εμείς θα θέλαμε να γίνεται αναφορά στη δίκαιη μετάβαση που θα διασφαλίζει ότι η κλιματική αλλαγή ε, συμβαδίζει με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και διασφαλίζει επίσης ότι οι βιομηχανίες μας κατευθύνονται προς ένα μέλλον με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα σε τομεακή βάση θέλουμε αυτό να ε, οδηγεί σε ένα οδικό χάρτη για το τι ακριβώς γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, όσον αφορά τώρα το θέμα των επιδοτήσεων, όπως σας είπα, είναι καλό να μειωθούν σιγά σιγά οι επιδοτήσεις που παρεμποδίζουν τη μετάβαση, αλλά το να συμπεριληφθούν οι λέξεις και οικονομικά επιζήμιες επιδοτήσεις. Εδώ τίθενται ερωτήματα τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε να υπάρχει μια κάποια μεγαλύτερη σαφάνεια. Και παρότι αναγνωρίζω ότι είναι σημαντικό για, την, για ε, ε, τις εκλογικές μας περιφέρειες να αναφέρουμε την ε, γεωργική βιομηχανία, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μια κάποια ανισορροπία στη γνωμοδότηση. Και ως προς τη μεταφορά τεχνολογίας, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δούμε ποια ακριβώς είναι η θέση του Κοινοβουλίου, να στηρίζουμε την τεχνολογία της επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, καλή συνεργασία, ε, ε, να υπάρχει ε, ανταλλαγή απόψεων στην επιστημονική δουλειά. Ένας από τους τομέες που λείπει είναι ο τομέας της ενεργειακής απόδοσης. Και αν δούμε λιγάκι τις τελευταίες εκθέσεις ε, από την IPCC ε, θα διαπιστώσουμε ότι επισημαίνεται η ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη ενεργειακή επάρκεια. Επάρκεια που άμεσα συνδεδεμένη με τα μοντέλα συμπεριφοράς. Ε, ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για περιορισμούς και αυτό θέλουμε να ενισχυθεί μέσα στην έκθεση. Επίσης, θα θέλαμε να προσθέσουμε να υπάρχει μια αναφορά ε, στη βιοενέργεια. Ε, η βιομάζα συνδέεται με την παγίδευση και την αποθήκευση του άνθρακα και αυτός είναι ένας τρόπος για να προωθήσουμε περαιτέρω αναφέρω τις ε, προτάσεις σε διεθνές επίπεδο. υπάρχει διεθνής διάλογος για την παγίδευση και την αποθήκευση του άνθρακα. Και πέρα από την ανάγκη τα κράτη να λάβουν μέτρα ε, οπουδήποτε μπορούμε πρέπει και διπλωματικά να διασφαλίζουμε ότι τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις που είναι απαραίτητες. Οφείλουμε να στηρίξουμε τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να προκύψει τελικά ε, περιορισμένη κατανάλωση του άνθρακα. Και τέλος, για να γίνουν όλα αυτά, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δέσμευση και ε, όσον αφορά στο ελάχιστο ποσοστό του ΑΕΠ που θα χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του άνθρακα. Εμείς προτείνουμε το 0,2% και αυτό ε, θα ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι όχι μόνο ηγούμεθα των κλιματικών ε, ενεργειών αλλά δεσμευόμεθα και οικονομικά στους προϋπολογισμούς μας. Ο Σνάλφος Πέντελε εκ μέρους ε, των φιλελευθέρων. Σα ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη για αυτή την γνωμοδότηση Μπορώ να συμφωνήσω επίσης ε, με τα περισσότερα πράγματα τα οποία είπατε κι εσείς και βλέπω ότι και οι παρατηρήσεις μας στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην γνωμοδότησή σας. Όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα όμως, είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή Ήτρε να αναφερθεί στο ζήτημα αυτό. Πρέπει όμως να καταφέρουμε να καταλήξουμε και στη σωστή διατύπωση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε έξυπνα το ζήτημα της διαρροής άνθρακα. Ξέρουμε ότι ο Επίτροπος Κανιέται θα κάνει μια παρουσίαση τον Ιούλιο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων και θα χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα benchmarking, συγκριτικής αξιολόγησης. Προφανώς εμείς λοιπόν πρέπει να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις αυτές που έχουν καλές επιδόσεις όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προσπίσουμε όμως με το νέο αυτό σύστημα και τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν καλές επιδόσεις. Ας μην τις προστατεύσουμε αυτές ενώ δεν θα έπρεπε στα πλαίσια του νέου ευρωπαϊκού συστήματο εμπορίας δικαιωμάτων. Ενδεχομένως να μην βασιστούμε αναγκαστικά στα αριθμητικά δεδομένα που έχουμε από το παρελθόν. Ξέρετε ότι για παράδειγμα ο τομέας της χαλιβουργίας παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως να ανακάμψει πάλι στο μέλλον. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ένα χάσμα, μία αναντιστοιχία ανάμεσα στο, στα δικαιώματα που θα έχει ο τομέας αυτός και στις πραγματικές του επιδόσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το benchmarking, το ζήτημα της, συγκριτι... της συγκριτικής αξιολόγησης. Όσον αφορά τώρα την βαθμία μείωση των επιδοτήσεων, συμφωνώ. Το πρόβλημα όμω είναι ότι όταν λέμε ότι οι επιδοτήσεις αυτές είναι επιζήμιες οικονομικά, τότε μπαίνουμε και σε μια οικονομική ιδεολογική συζήτηση για το τι είναι επιζήμιο και τι δεν είναι. Εγώ ως φιλελεύθερος θα έλεγα ότι οποιαδήποτε επιδότηση είναι οικονομικά επιζήμια, άλλοι πάλι μπορούν να διαφωνούν με αυτή την άποψη. Σε κάθε πάντως περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις περιβαλλοντικά επιζήμιες επιδοτήσεις. Η υφιστάμενη πάντως διατύπωση δεν ξέρω αν μας καλύπτει. Χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή επιδοτήσεων για ορεικτά κάψιμα στην Ευρώπη, για πετρέλαιο και άνθρακα. Τα χρήματα αυτά θα είχαν πολύ καλύτερη χρήση σε άλλους τομείς. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο, αν προβλέπαμε τέτοιες μειώσεις των επιδοτήσεων, θα προετοιμαζόμασταν καλύτερα και για τη συνδιάσκεψη των Παρισίων. Νομίζω πάντως ότι έχουμε ξεκινήσει καλά και ότι υπάρχει τώρα μια στοιχειώδη θετική ε, συνεννόηση ανάμεσα σε όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει τώρα να καταλήξουμε σε έναν επικοδομητικό συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Ζαντό τώρα έχει το λόγο εξ των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συντάκτη γνωμοδότηση Οι συνάδελφοί μου οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι ήδη με κάλυψαν εν μέρη. Προφανώς θα πρέπει να δώσουμε μία μάχη, μία μάχη κατά της διαρροής άνθρακα. Ανέκαθεν λέγαμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύσει τις βιομηχανίες από τις οποίες ε, ζητούμε να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες και οι οποίες ε, καταβάλλοντας προσπάθειες αυτές απειλούνται από το λεγόμενο κλιματικό dumping. Τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι η βιομηχανική κλάδη εκείνη που απειλούνταν περισσότερο από τον εξωτερικό ανταγωνισμό είναι η κλάδη εκείνοι οι οποίοι αποφελήθηκαν τελικά περισσότερο από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων καθότι έχουν καταφέρει να εξοικονομήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, πολλές φορές και ένα δισεκατομμύριο ευρώ, όπως για παράδειγμα η Arcelor μέσω του ευρωπαϊκού ETS κατάφεραν κατά αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουν ε, ένα πολύ σημαντικό αριθμό δικαιωμάτων εκπομπών. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ποιους προστατεύουμε και πόσους προστατεύουμε. Επίσης, το όλο ύφος της έκθεσης αυτής δίνει την εντύπωση αφενός και αυτό είναι θετικό ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το κλίμα. Από την άλλη όμως χρειάζεται και μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή ηγεσία όσον αφορά τον ε, μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Καλόν το κάνουμε αυτό, αλλά θα πρέπει και οι υπόλοιποι να κάνουν κάτι τέτοιο διαβάζοντας τις εκθέσεις ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ενέργειας, διαβάζοντας τελευταία έκθεση για την, από την Ιρένα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις Ανώσιμες Πηγές Ενέργειας, βλέπουμε ότι αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τον επενδύσει κανείς και στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις ανανεώσιμες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, πολλές φορές καταφέρνουν χωρίς καμία επιδότηση να έχουν τελικά το ίδιο κόστος με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και αν συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μας λέει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα ορυκτά καύσιμα δέχονται ως επιδοτήσεις 10 δισεκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια ευρώ κάθε λεπτό. 5,3 δισεκατομμύρια σε τήσια βάση πηγαίνουν ως επενδύσεις στα ορυκτικά καύσιμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν λάβετε υπόψη στα στοιχεία αυτά, ότι πραγματικά αξίζει τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την απασχόληση να κινηθούμε όλο και περισσότερο προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρουμε ότι δεν θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε διεθνή συμφωνία στο Παρίσι, αν η ίδια η Ευρώπη δεν αναλάβει ηγετικό ρόλο, δεν είναι οι Κινέζοι ούτε οι Αμερικάνοι αυτοί που θα αναλάβουν τέτοιο ηγετικό ρόλο σε μια τέτοια διεθνή διάσκεψη. Είναι η Ευρώπη αυτή που πρέπει να αναλάβει τα ενία, αλλά δεν θα πρέπει να είναι μόνο φιλόδοξη όσον αφορά τη διάρθρωση που θα έχει αυτή η συμφωνία. Θα πρέπει παράλληλα η Ευρώπη να έχει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τον βιομηχανικό, ενεργειακό, γεωργικό, μεταφορικό μετασχηματισμό. Αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν οι πόλεις και οι περιφέρειες στην Ευρώπη. Αν δείτε για παράδειγμα την έκθεση από την Σύμβαση των Δημάρχων, αυτό το οποίο γίνεται ήδη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ δυναμικό. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό κοινοτικό επίπεδο δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε τη δυναμικότητα, την ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι περιφέρειες και οι τοπικοί παράγοντες στην Ευρώπη. Ας μην λοιπόν υποχωρήσουμε μπροστά σε κάποια συμφέροντα τα οποία τελικά έχουν ως στόχο να επιβραδύνουν τον ενεργειακό μετασχηματισμό στην Ευρώπη και κατά αυτόν τον τρόπο επιβραδύνεται και οποιαδήποτε ελπίδα της Ευρώπης να κατευθυνθεί προς μια οικονομική ανάκαμψη. Ας είμαστε λοιπόν εμείς στην ε, σωστή πλευρά, αν θέλετε, των πραγμάτων, α συνταχθούμε περισσότερο με εκείνου οι οποίοι προωθούν τι νέε μορφέ ενέργεια για τον 21ο αιώνα. Και επιτέλου α σταματήσουμε να λέμε Μα εμεί δεν κάνουμε τίποτα ή α μην κάνουμε τίποτα τη στιγμή που οι Καναδοί, οι Αυστραλοί, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι δεν κάνουν τίποτα. Δεν θα καταλήξουμε ποτέ σε τίποτα το θετικό αν υιοθετούμε τέτοια στάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. συνάδελφο Φερέιρα, εκ μέρου ε, τη ε, ΓΚΟΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω αρκετά πράγματα που θα μπορούσα να αναφέρω. Καταρχήν όσον αφορά το σχέδιο για το οποίο συζητάμε και όσον αφορά και όλα τα άλλα τα οποία μόλις τώρα ανέφεραν συνάδελφοι. Θα είχα λοιπόν πάρα πολλά να πω αλλά δεν θα τα πω γιατί πιστεύω ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η συζήτηση διότι μέχρι πριν από 10 λεπτά είχαν γίνει μεταφράσει σε 6 μόνο γλώσσες. Λιγότερο δηλαδή από το 1 τρίτο των επίσημων ε, γλωσσών ε, στις οποίες ε, θα έπρεπε να έχει υποβληθεί το ψήφισμα. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, στη δική μου την έκθεση παρεπιπτόντος για την μπλε οικονομία, επί της οποίας μόλις πριν από λίγο ψηφίσαμε, και εκεί συνέβη ακριβώς το ίδιο. Και εγώ είχα αρνηθεί να γίνει η συζήτηση αν δεν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες μεταφράσεις. Νομίζω λοιπόν ότι όλες οι πολιτικές ομάδες ε, θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Κοιτάξτε, αυτό πια δεν είναι εξαίρεση. Κανόνας έχει γίνει. Και κατ' ουσίαν εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι ισχύει η αρχή της πολυγλωσίας και την πολυγλωσία δεν μπορούμε να την αγνοούμε. Αυτό είναι ακρογωνιαίος λήθος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν, τέλος, εγώ δεν συζητώ, αρνούμε. Και σε το λέω αυτό εκφράζοντας τη βαθιά μου λύπη είναι μια διαμαρτυρία αυτή εκ μου και σας παρακαλώ πολύ απευθύνω έκλεισε όλους να το σκεφτούν σοβαρά το θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι έχουν γίνει αποφάσεις, έχουν αποφάσεις να γίνουν περικοπές και στη μετάφραση και στη διερμηνία και πρέπει να σκεφτούμε αυτό πώς θα πειράσει τη δουλειά μου. Γιατί σας λέω, επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια ακρογωνία, ε, έναν ακρογωνιαίο λίθο ε, της δουλειάς μας που είναι η πολυγλωσία. Έκκληση είναι αυτή που απευθύνω, λυπάμαι πάρα πολύ, διαμαρτύρομαι. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να γίνει γρήγορα μετάφραση και αυτό σημαίνει συχνά, έχει τα λεφτά το κοινοβούλιο να πληρώσει. Να πληρώσει, να μεταφράσει, να γίνει διερμηνία, έτσι πρέπει να γίνεται. Uh, Πρόεδρος, έχετε δίκιο ότι η πολυγλωσία είναι καθοριστική ε, συμφων... σημασίας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποτελείται από 28 κράτη-μέλη και από 24 γλώσσες που είναι επίσημες γλώσσες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν επίσης και οι κανονισμοί. Το έχετε αναφέρει αυτό ήδη κάνα δυο φορές κατά το παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι για να γίνει ψηφοφορία χρειαζόμαστε ε, όλες τις μεταφράσεις. Βεβαίως ε, αυτό λυπάμαι πάρα πολύ δεν ισχύει για τη συζήτηση, ισχύει για την ψηφορία. Εντάξει, ε, δεν είναι βέβαια... Δεν σημαίνει ότι κακώς κάνατε που μας τα υπενθυμίσατε γιατί μπορούμε να αλλάξουμε τους ε, κανόνες. Γι' αυτό βέβαια είναι αρμόδια επιτροπή ΑΦΚΟ. και μπορούμε να τους διαβιβάσουμε την πρόταση, αλλά τώρα η διαδικασία είναι αρκετά σαφής. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάστηκαν να σας τα πω αυτά που σας είπα. Σαφώς και είναι καλό για όλους μας ε, να έχουμε τις μεταφράσεις. Να το υπογραμμίσω αυτό ότι όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά για μας. Σας ε, στηρίζω, αλλά όπως σας είπα έχουμε και τους δικούς μας τους κανόνες και δεν είναι πάντα ε, δυνατό να έχουμε όλες τις μεταφράσεις για τη συζήτηση. Λυπάμαι πάρα πολύ και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε. Στο τέλος υπάρχουν όλες οι μεταφράσεις. Αυτές θα είναι έτοιμες για να μπορούμε να ψηφίσουμε. Ε, από αυτό δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς να υπάρχουν μεταφράσεις και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέλλον. ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις. Παρακαλώ, η συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ που με έχετε βάσει στην κατηγορία λύπη ομιλητέ. Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή η γνωμοδότησή του νομίζω ότι είναι μια καλή βάση για να αναπτύξουμε ακόμη περαιτέρω το θέμα. Θέλουμε να δούμε τα πιο προεξέχοντα ζητήματα αναφερόμενοι και στην ανταγωνιστικότητα. Είναι ωραία όμως ε, η ε, κατεύθυνση ότι πιστεύω ότι ο στόχος μας στο Παρίσι θα πρέπει να είναι η δεσμευτική στόχη από όλε τι μεγάλε χώρε για να αντιμετωπίσουμε τα πρόβλημα τη θεωρή άνθρακα και για να προχωρήσουμε σε νέε αποδοτικέ ω προ το κόστο μειώσει. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει ότι όλε οι χώρε στη Συμφωνία Αλλαγή του Κλίματο ε, θα μπορούν να τηρήσουν τι δεσμεύσει του. Τέλο, όπω προπόθηκε, θα πρέπει όπου χρειάζεται να δίνεται υποστήριξη, αλλά κάθε χώρα να είναι η πόλη σε μη συμμόρφωση. Επίση, η αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα είναι σημαντική για να αντιμετωπίσουμε ορθά το πρόβλημα τη αλλαγή του κλίματο. Το λέει και η γνωμοδότηση. Και σε ό,τι αφορά το αποθεματικό σταθερό τη αγορά, καλό είναι αυτό. Αλλά δεν είναι και τόσο σαφέ αν θα διορθωθεί με τον τρόπο αυτό η δομική, ε, το δομικό πρόβλημα του ETS Θέλουμε να έχουμε αποδοτικότητα του κόστους και να μην έχουμε απλά και μόνο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, γιατί θα έχουμε διευρύνει τις ενεργειακές πηγές. Και κάτι άλλο που είδα είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ αλλαγής του κλίματος και θαλάσσου περιβάλλοντος και πράσινη οικονομία. Επίσης, οι μεταφορές που είναι μετά την ενέργεια υπεύθυνε για το μεγαλύτερο ε, μερίδιο εκπομπής, άνθρακ. Θα έλεγα ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο διεθνές επίπεδο νέες πολιτικές που δεν θα περιοριστούν στα εθνικά γεωγραφικά σύνορα για περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Σε αυτά θα κινηθώ στην, ε, στις μου. Ε, I understand Σταμπουράνο νομίζω ότι θέλει το λόγο και μέρος της ομάδας EFTD. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που στην γνωμοδότηση αυτή βλέπουμε ότι όντως στρεβλώνεται η εσωτερική αγορά από τις επιδοτήσεις που δίνονται στα ορυκτά καύσιμα. Βασιζόμαστε επίσης σε μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μας λένε ότι οι άμεσες αυτές επιδόσεις που δίνονται προς τα ορυκτικά καύσιμα έχουν φτάσει τα 5.000 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι δυστυχούν σε ένα τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ οι επιδοτήσει αυτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα σε οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο από επιστημονικής πλευράς. Μολονότι αυτή τη στιγμή λέμε ότι θα θέλουμε να προωθήσουμε τις προτεραιότητες της ΣΥΤΡΕΣ, πρέπει να δούμε επίσης και ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα. Σε αυτά δυστυχώς δεν αναφερόμαστε στην έκθεση αυτή. Στην παράγραφο 5 νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι η ανάλυση που έχουμε εδώ πέρα ουσιαστικά έχει την ευρύτερη υποστήριξη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Αν θέλουμε πραγματικά να δείξουμε ότι υπάρχει επιστημονική διασύνδεση ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και τη διατήρηση της βιωσιμότητος, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι κλιματικές αλλαγές έχουν αρχίσει να έχουν βιομηχανικές και περιβαλλοντικές όμως επιπτώσεις. Στην παράγραφο 7 της έκθεσης του κυρίου Κέλλη υπάρχει η εξής φράση «Υπογραμμίζει τις, τα οικονομικά ωφέλη που μπορούν να προέλθουν για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ουσιαστικά ναι, να λέμε εδώ πέρα «Υπογράψτε τις συμφωνίες και εμεί θα καταφέρουμε να καρποθούμε όλα τα ωφέλη» από οικονομικής πλευράς αναφερόμαστε μόνο στην κλασική οικονομία, στον κλασικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Νομίζω θα πρέπει ανταυτού να αφαιρθούμε περισσότερο στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες, οι οποίες συμβάλλουν στην ευημερία της κοινωνίας. Τέλος, να καταλήξουμε την εξής παρατήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα ενέκρινε ένα ψήφισμα που είναι ιδιαίτερα συντηρητικό κατά την άποψή μας ε, όσον αφορά το 2% του ΑΕΠ των κρατών μελών που μπορεί να δοθεί στις αμυντικές βιομηχανίες. Αν ο πραγματικός εχθρός όμως της ανθρωπότητας είναι πλέον τον αιώνα αυτό οι κλιματικές αλλαγές, τότε νομίζω θα ήταν πολύ πιο σόφρον να δίνουμε χρήματα από το Εθνικό ΑΕΠ για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε τελικά σε οικονομίες και κοινωνίες με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κάθλιν Βαν Μπρέντ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ γρήγορα να πω για τους μόνο τους συναδέλφου. Μία σημαντική αποστολή που έχουμε ως πολιτική είναι να πείθουμε την κοινή γνώμη Καλή είδηση λοιπόν στο μέτωπο αυτό είναι ότι αυτήν την εβδομάδα μπορεί να ακούγεται περίεργο αλλά δεν είναι ότι πρώτη τελευταία φορά ο Πάπας που είναι ιδιαίτερος και το λέω αν και δεν είμαι καθολική έτσι αυτήν την εβδομάδα λοιπόν μια παπική εγκύκλειος ε, που κυκλοφόρησε αναφέρεται στην αλλαγή του κλίματος, τη φτώχεια, την οικονομία, την κοινωνία. Εγώ πιστεύω πολύ στις τεχνολογικές λύσεις και πιστεύω ότι μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα, αλλά πρέπει να μπορούμε να πείθουμε και ε, τον κόσμο. Να αγγίξουμε την καρδιά των ανθρώπων πρέπει να κάνουμε και αυτό το κάνει ο Πάπας πιστεύω. Και ακούγεται και ότι η συντηρητική Αμερικανία είναι πολύ αρνητική ως προς το κλίμα. Τώρα, έρχομαι στο δεύτερο, G7. Σε ό,τι αφορά τους δύο βαθμούς Κελσίου. Και εκεί υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Ε, τώρα εμείς, σε ό,τι αφορά τις μέρες μας, δεν μπορούμε να τους υποστηρίξουμε. Γιατί αν πετύχουμε τις δεσμεύσεις μας, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3,5 και κατά 4 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Άρα πρέπει οι στόχοι μας να βελτιωθούν. Θα πρέπει να ορίσουμε μια καλή μέθοδο. Να εξεύρουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και να έχουμε και ηγετική στάση. Ελπίζω, γιατί βασίζομαι και στον σκιώδη των συντάξεων νομοδότηση, για την εξέβρεση μιας καλή συμφωνία. Και ελπίζω η Ήτρε να μην παραμείνει σιωπηλή, αλλά να γίνει ακουστή η φωνή και η άποψή μα. αφού και ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι είναι σημαντικό το κλίμα για την ανθρωπότητα, έχουμε επιχειρήματα. Ίσως να ήταν και μια αναμενόμενη δήλωση αυτή, αλλά πολύ σημαντική Κάριντς. Σας ευχαριστώ πολύ. Άκουσα όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κέλλη για την ε, ισορροπημένη αυτή γνωμοδότηση. Αλλά θα ευχόμουν πραγματικά στην Ευρώπη να αντιστοιχούσαμε σε διαφορετικό ποσοστό και όχι σε αυτό το 11% των εκπομπών Λέμε ότι στην Ευρώπη πρέπει να σταματήσουμε την τάση αυτή, αλλά εμεί ελέγχουμε τελικά μόνο το 11% των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ακόμα και να μηδενίσουμε αυτέ οι εκπομπέ δεν πρόκειται να σώσουμε τον πλανήτη, αν αυτό είναι ο στόχο μα. Συνεπώ, θα πρέπει να καταφέρουμε να πείσουμε του εταίρου μα στι ΗΠΑ και την Κίνα κυρίω, αλλά και την Ινδία, να αναλάβουν δράση και ουσιαστικά να ακολουθήσουν τις ιδέες αυτές που τόσο εύκολα αποδεχόμαστε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Πρόσφατα ήμουνα σε ένα δείπνο μαζί με νομοθέτες βουλευτές από την Επιτροπή Ενέργειας της Αμερικής και συζητούσαμε μαζί τους 3-40 λεπτά και ένας ο οποίος είναι από τους δημοκρατικούς, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τους δημοκρατικούς σοσιαλιστές αριστερούς, διέκοψε τη συζήτηση και είπε μια στιγμή, μα δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι δεν καταλαβαίνετε, του είπαμε, Πώ το διάλογο, νομίζω ότι χρησιμοποίησε τη φράση αυτή, πώ θα εξηγήσετε στου ψηφοφόρου σα ότι οι ψηλότερες τιμέ ενέργεια είναι κάτι το θετικό. Και εγώ το απάντησα, μα κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Είπα ότι βασική μας, ο βασικό μα στόχο είναι να μειώσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό μου απάντησε, μα θα ήσασταν νεκρός, θα σας σταύρωναν στι Ηνωμένε Πολιτείε, αν κάνετε κάτι τέτοιο. Για τις Ηνωμένε Πολιτείε, τον τελευταίο λόγο είχε ανταγωνισμό, ανταγωνιστικότητα. Η δυσκολία λοιπόν αυτή τη στιγμή έγκυται στο ότι στη συζήτηση που κάνουμε δεν υπάρχει καμία σύγκριση όσον αφορά τις τιμές, δεν γίνεται συζήτηση όσον αφορά τις τιμές τη ενέργειας. Γιατί εμείς τελικά μπορεί να καταλήξουμε στο να εξαλείψουμε εντελώ τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα καταφέρουμε ακόμα και τότε να σώσουμε τον πλανήτη, αν οι εταίροι μας δεν αλλάξουν συμπεριφορά. Οι στόχοι που θέτουμε λοιπόν στην έκθεση αυτή είναι στόχοι που γίνονται γενικότερα αποδεκτοί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με κάποιες μεμονωμένε βέβαια εξαιρεσει που δεν πιστεύουν φαντάζομαι στα επιστημονικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε ανταυτού όχι μία ευρωπαϊκή συμφωνία, αλλά μία παγκόσμια συμφωνία. Τι θα κάνουμε όμως απουσία τέτοια συμφωνίας. Μπορούμε πραγματικά εμείς να γίνουμε ουραγοί της όλης διαδικασίας. Εγώ προέρχομαι από τη Λετωνία, μια χώρα ιδιαίτερα πράσινη. Το 1 τρίτο της ενέργειάς μας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θεωρώ ότι θέτουμε αυτή τη στιγμή ένα θεαματικό παράδειγμα. Ο λόγος ενδεχομένως είναι το ότι δεν έχουμε ένα πολύ ανεπτυγμένο βιομηχανικό τομέα. Ενδεχομένως γι' αυτό να ευθύνει το ότι είχαμε για 50 χρόνια σοβιετική κατοχή. Τώρα, στόχος μας είναι να γίνουμε όλοι οικολόγοι, πράσινοι και φτωχοί συνάμα, δεν ξέρω. Συνεπώς κάνω τις παρατηρήσεις αυτές και εκφράζω κάποιες πρώτες ιδέες γιατί καταλαβαίνω ότι πολύ συχνά είμαι μόνος μου στην όλη αυτή συζήτηση, είμαι λίγο αποκομμένος αυτή την όλη συζήτηση. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή και θα ήθελα αυτό ενδεχομένω να το σχολιάσουν και οι συνάδελφοι, είναι ότι ο κόσμο δεν απαρτίζεται μόνο από πολιτικού, αλλά από βιομηχανίε και σε άλλε χώρε οι οποίε βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με την Ευρώπη. Τι κάνουμε λοιπόν εμεί για αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει. Δεν λέω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, δεν στρέφομαι κατά των επιστημονικών δεδομένων. Το μόνο το οποίο λέω είναι πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε και τις υπόλοιπες οικονομίες ότι πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μας το παράδειγμα. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε έχουμε λύσει και το πρόβλημα. Έχετε και μία μπλε κάρτα, μία μπλε κάρτα από τον κύριο Ζαντό. Δεν έχουμε μπλε κάρτες, αλλά έχω και πολλή φαντασία. Δεν είναι ακόμα πράσινη κάρτα. Ε, κοιτάξτε, Ακούστε. Για το Σάφο η μετάβαση, ε, η ενεργειακή μετάβαση δεν ε, θα συζητηθεί μόνο στο Παρίσι. Αν δει κανεί εκθέσει ε, που δημοσιεύονται και δει κανεί και τι οικονομικέ αναλύσει ότι αυτό το κόστο των διαφόρων πηγών ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, εδραυλική βιομάζα υδροελεκτρική, αιωλική κτλ. Το κόστος παραγωγή σήμερα είναι σχεδόν ισοδύναμο με το κόστο των ορκτών καυσίμων και τη ε, πυρηνική ενέργεια. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Δεν το λέει η οικολογία, δεν ε, είναι ε, η δική μας σκιαμαχία, να σκοτώσουμε τη βιομηχανία και αυτό το βλέπουμε, το διαβάζουμε τις εκθέσεις. Για ένα εκατομμύριο ευρώ που επενδύεται στις διάφορες πηγές ενέργειας Έχουμε 1,5, 1,5 θέσεις εργασίας ε, στα ορυκτά, καύσιμα, μια μισή στον πυρηνικό τομέα. Η ολική ενέργεια στη Γερμανία είναι 7 θέσεις εργασίας. Εκεί είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ένα έλλειμμα ε, πληροφόρησης στο πώς θα ενημερώσουμε τους πολίτες. Ε, πέρασε ο χρόνος σας. Πρέπει να είμαστε λογικοί σήμερα, αυτοθολογιστές. Ευχαριστώ κύριο Φέντριλε. Δεύτερη μπλε κάρτα Ναι, ξέχασα να πω κάτι στον κύριο Κέλλη. Για το copyright, τα δικαιώματα δημιουργού, δεν θα πρέπει να κλιμακωθεί ο πόλεμος που γίνεται στο Κοινοβούλιο για τη μεταρρύθμιση τη σχετική νομοθεσία. Σίγουρα πρέπει να προστατεύσουμε τα πνευματικά δικαιώματα τη ε, ε, βιομηχανία, αλλά να μην δημιουργήσουμε ε, πολιτικό μπάχαλο, αν μου επιτρέπετε. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Κάριν στη Σουηδία έχουμε πολύ ψηλό φόρο ε, του άνθρακα. Συν το σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Αλλά η βιομηχανία μα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική από άλλε χώρε. Έχουμε χαμηλότερε εκπομπέ και όταν έρχεται το τιμολόγιο ε, του ρεύματο και σε μένα και στη βιομηχανία είναι πολύ χαμηλότερο. Και αυτό οφείλεται στο ότι λειτουργεί αγορά. Το πρόβλημα ίσω είναι εκεί δεν ξέρω τι γίνεται στην Εστονία, ε, πρέπει να δημιουργούμε πάντως ε, αγορές που να λειτουργούν σωστά, γιατί αυτό μειώνει και τις τιμές. Αν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή, να μην υπονομεύσουμε τον ηγετικό ρόλο της Ένωσης για να έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία, πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια ισχυρή θέση. Αν δεν έχουμε ισχυρή θέση, θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Μην ξεκινήσουμε από αυτό, για να μην υπονομεύσουν από μόνοι μας τη θέση μας. Ευχαριστώ πολύ, πέρασε ο χρόνος σας. Κριστιανής, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το λόγο. Κάνω όλα ξεκάθαρα στη συζήτηση. Κάρνη, συμφωνώ απόλυτα ότι οι αγορές και οι τιμές είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για τις αλλαγές που θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Αξιοτιμότατε, κύριε επικεφαλής των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Κλίμα. Κύριε Μέτσγκερ, έχετε το λόγο. Thank uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε δυνατότητα στην Επιτροπή να πει και αυτή λίγα λόγια. Νομίζω λοιπόν ότι από τη συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε ότι στηρίζουμε πλήρως ε, την άποψη της Επιτροπής Ήτρε. Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Επίσης ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για το ότι ε, θέλουμε να βρεθεί μια λύση για τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων λόγω διαρών του άνθρακα. Και επίσης ε, θέλω να πω ότι μας ενδιαφέρει όλες οι μεγάλες οικονομίες να καταστούν μέλη και να υπογράψουν τη Συμφωνία των Παρισίων. Αν ληφθεί η απόφαση στο Παρίσι, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει επικύρωση αυτή της συμφωνίας και αυτό σημαίνει ότι όλοι από τους 196 ε, διαπραγματευτές θα πρέπει να επανέλθουν στα κοινοβούλια τους για να ζητήσουν την επικύρωση. Άρα δηλαδή το Παρίσι δεν είναι το τέλος της συμμετοχής του Κοινοβουλίου. Θα υπάρξει αναμφισβήτητα μετά το Παρίσι άλλη μια ευκαιρία για να συζητήσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις για την οικονομία. Τώρα, όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, ο πρόεδρος κύριος Γιούγκερ επιθυμεί ε, να δρέψει τα αποτελέσματα την αμέσως επόμενη δεκαετία για να διασφαλίσει τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και θέλει επίσης ε, να παραμείνουμε ε, πρωτοπόροι, ε, η κορυφή, η αιχμή του δόρατος θα έλεγα ε, όσον αφορά τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες διότι αυτές που έχουν ανάγκη βέβαια μπορεί να μην έχουν ανάγκη όλες μπορούμε και να προσφέρουμε και την τεχνική μας υποστήριξη που έχουμε από την εμπειρία μας μετά την εφαρμογή ενεργειακών πολιτικών στην Ευρώπη. Ε, σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Η Κίνα εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά ε, την, ε, το κλίμα, άρα δηλαδή όλα αυτά δεν έχουν σχέση μόνο με το κλίμα και σε διμερές επίπεδο πρέπει να λάβουν χώρα διαπραγματεύσεις για να πείσουμε τους εταίρους μας. Με τις ΗΠΑ και την Κίνα είμαστε ιδιαίτερα επιτυχεί στις τελευταίες δεκαετίες. Χρειαστήκαμε αρκετό καιρό για να συμπεριλάβουμε και αυτές τις χώρες και νομίζω προς το παρόν τουλάχιστον όλα αυτά πολύ σωστά συμπεριλαμβάνονται στις ε, προτάσεις μας. Και οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί στο να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα εφέτος στο Παρίσι στις διαπραγματεύσεις. Με αυτά λοιπόν ολοκληρώνω την παρέμβασή μου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Μα και εμεί σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν παρόν και που ακούσατε όλη αυτή τη συζήτηση. Ο κύριο Σον Κέλλη, το αρχιτολόγο, ο συντάκτη γνωμοδότησης, θέλετε να πάρετε το λόγο για πόσο, ένα λεπτό ή για περισσότερα λεπτά. Όχι για πολύ χρόνο κύριε Πρόεδρε, δεν θα με ακρηγορήσω. Θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω του συναδέλφου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι παρατήρησει του εν γέννη. Νομίζω ότι έχουμε πλέον μία βάση για μία καλή έκθεση Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαμε με τα βασικά σημεία της έκθεσης αυτής να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις μόνο. Όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση, το benchmarking, τις επιδοτήσεις, την ενεργειακή αποδοτικότητα, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να γίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της καινοτομίας πολύ πιο ελκυστική στο μέλλον. Ξέρετε ότι πριν από δύο εβδομάδε διάβασα μια πάρα πολύ καλή έρευνα που είχε να κάνει με μια νέα μορφή ενέργεια, την παλιριακή ενέργεια. Νομίζω ότι και αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει πολύ στο πεδίο ε, ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει προφανώς να ασχοληθούμε και με την ίδια την ε, γεωργική πολιτική και να δούμε πώς διασυνδέεται με την κλιματική αλλαγή και πώς επηρεάζει τελικά την επιστηστική ασφάλεια. Επίσης πρέπει να συνδέσουμε τις προτάσεις αυτές και με το πρόβλημα της αποψήλωσης των δασών σε ορισμένες χώρες. Όσον αφορά τώρα τις, τα σχόλια του κύριου Κάρενς, είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε μια δεσμευτική συμφωνία, αλλά ποια θα είναι η τακτική μας. Θα πάμε στο Παρίσι και θα πούμε ότι ανεξάρτητα με οτιδήποτε γίνεται εδώ πέρα, εμείς θέτουμε αυτούς τους στόχους ή θα πούμε, κοιτάξτε, είμαστε έτοιμοι να συμβαστούμε, αλλά θα πρέπει και εσείς να κάνετε κάποιε υποχωρήσει και αν δεν κάνετε υποχωρήσει θα αναθεωρήσουμε και εμεί τη στάση μα. Είναι θέμα τακτική. Πρέπει να θέσουμε προφανώ στόχου, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποια καθεστώτα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα δημοκρατικά. Ξέρω ότι πολλές φορές οι συζητήσεις αυτές συμμετέχουν ακόμα και κάποια αυταρχικά καθεστώτα. Όλοι με τον έναν άλλο τρόπο θα πρέπει να καταφέρουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία στο Παρίσι. Και αν καταλήξουμε στην παγκόσμια αυτή συμφωνία θα σώσουμε τον κόσμο, αν όχι δεν θα σώσουμε τον πλανήτη. Και τότε τι κάνουμε. Και ξέρετε ότι ε, η Κίνα, η οποία αντιστοιχεί στο 25% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, ο οποίο πρέπει και αυτός να κινηθεί προς τη δική μα την πλευρά. Σα ευχαριστώ πολύ πάντως, σας ευχαριστώ πολύ για τι παρατηρήσει σα, Πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τις τροπολογίες για αυτή την γνωμοδότηση, 30 Ιουνίου 2015, 12 το μεσημέρι είναι η καταληκτική προθεσμία. Σε δύο εβδομάδες περίπου. Και στη συνέχεια θα γίνει η ψηφοφορία στην Ήτρε, στην Επιτροπή μας, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το πιο σημαντικό πάντως να θυμάστε ότι η καταληκτική προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι η 30 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Θα σας δω πάλι στις 3 το μεσημέρι για το τελευταίο τμήμα της συνεδρίασής μας. Για 3,5 ώρες θα συνεδριάσουμε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ.